Παρακαλώ καθίστε για να ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα της εκλογής. Εψήφισα 729, άκυρα 12, έγκυρα 717 ψηφοδέλτια. Αυτό σημαίνει ότι η απόλυτη πλειοψηφία είναι 359 ψήφους. Σας διαβάζω με αλφαβητική σειρά. έλαβων. Καστάλτο. 113 ψήφους. Η κυρία Κρέτσου. 442. Τσερνέτσκι. 240. Η κυρία Γκάλ 400. Η κυρία Γκυγιόμ 334. Ο κύριος Λάμστροφ 311. Η κυρία Λούνατσεκ 222. Η κυρία Μαγκίνες 441. Ο κύριος Παπαδημούλης 153. Ο κύριος Ρεν 327. Ο κύριος Σασόλη 340. Ο κύριος Σταγιάννη, 452. Ο κύριος Βαλκάρσελ Σίσο. 406. Η κυρία Βαλεάν. 394. Και ο κύριος Βίλαντ 437 ψήφους. Η απόλυτη πλειοψηφία έχει καλύφθει από τον κύριο Ταγιάννη, την κυρία Μαγκίνες, τον κύριο Βίλαντ, τον κύριο Βαλκάλσερ Σιζό, την κυρία Γκάλ Πέλτς και την κυρία Βαλεάν. Συγχαρητήρια προς τους συναδέλφους αυτούς που ήδη εξελέγησαν. Αυτό τώρα τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να καλυφθούν άλλες 8 θέσεις αντιπροέδρων και θα ακολουθήσει δεύτερος γύρος εκλογών. Εάν δεν υπάρχουν σχόλια, θεωρώ ότι οι υποψήφοι και οι υποψήφιες του πρώτου γύρου διατηρούν την υποψηφιότητά τους. Δεν αποσύρεται κανείς. Δεν βλέπω καμία αντίρρηση διαφωνία. Ισχύουν λοιπόν οι υποψηφιότητες και προτείνω να προβούμε τώρα στη δεύτερη εκλογή στο δεύτερο γύρο. κύριος Βέμπερ, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να παρακαλέσω να κάνουμε μια σύντομη διακοπή ενό δεκαλέπτου για να έχουμε κάποιες διαβουλεύσεις στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και άλλες ε, για να δούμε ε, πώς θα χειριστούμε το αποτέλεσμα. Εάν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, παρακαλώ. Ο Πρόεδρος, προτείνω μικρή διακοπή μέχρι τις 5 και 20. Διακόπτε τη συνεδρίαση.